Wznawiam posiedzenie. Protokół z wczorajszego posiedzenia. Συνεχίζεται η συνεδρία. Τα χθεσινά πρακτικά έχουν ε, διανεμηθεί. Υπάρχουν σχόλια, φαίνεται πως όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι τα χθεσινά πρακτικά έχουν εγκριθεί. Η ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα προβλέπει μια κοινή συζήτηση τεσσάρων εκθέσεων που σχετίζονται με το θαλάσσιο πακέτο και θα δώσουμε το λόγο καταρχήν στον ε, κύριο Ντεγκράντες Πασκουάλ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Ταγιάννη, κυρίες και κύριοι, σήμερα